Good afternoon, dear colleagues. And welcome to... Και καλώς ορίσατε στην πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Κυρίσω την έναξη της συνεδρίασης και θα ήθελα να ξεκινήσω ε, με συγχαρητήρια προς όλους σας ε, για την εκλογή σας, την επανεκλογή σας σε πολλές περιπτώσεις. Να σας συγχαρώ επίσης για την απόφαση να έλθετε να εργαστείτε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, μία από τις πλέον σημαντικές επιτροπές του Κοινοβουλίου, η οποία από την πρώτη μέρα θα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για τον μελλοντικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027 και σας εύχομαι και πάλι λοιπόν ε, καλή αρχή. Θα προεδρεύσω στο πρώτο τμήμα της συνεδρίασης. Είμαι αυτό που λέμε μεταβατικός πρόεδρος για να επιτελέσω χρέη προέδρου στην εκλογή του πρόεδρου. Και μοναδικό σκοπό τη σημερινή μα συνεδρίαση, συνάδελφοι, είναι να εκλέξουμε τον πρόεδρο τη Επιτροπή και του τέσσερι αντιπροέδρου. Τι θα κάνουμε λοιπόν, Καταρχά θα εκλέξουμε προφανώ τον πρόεδρο και μετά τους τέσσερις αντιπροέδρους. Τα μέλη της Επιτροπής να έχουν ε, υπόψη του ότι χρειαζόμαστε κάρτες για την ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Αν δεν έχετε παρακαλώ τις κάρτες σας, ζητήστε από τους βοηθού σας να πάρουν μια κάρτα από τον τρίτο όροφο. Στη συνέχεια, να σας ενημερώσω για το ποιοι είναι οι αναπληρωματικοί που αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη. Ο Ματέν Ντενεόλφη, την αναποβρίσκω αντικαθιστά, η Κλέρ Φόξ, τον Τζόναθαν Μπόρακ, αναλύσα τον Βαλεντίνο Γκοάν, ο Μάριο Φορόρε, τον Ρούπερτ Λόου, η Μελέτα Αλελούτσι, τον Ένικα Νίλσεν και ο κύριο Ντόρφμαν, τον κύριο Βίλαντ. Αν έχουμε και άλλους αναπληρωματικούς που αντικαθιστούν τακτικά μέλη, σας παρακαλώ ενημερώστε τη γραμματεία. Πριν την έναξη της ε, ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στην ε, εκλογή του νέου Προέδρου. Καταρχάς, να δούμε κατά πόσον έχουμε απαρτία. 41 μέλη, χρειαζόμαστε 11 μέλη για την απαρτία και έχουμε παρόντα παραπάνω από 11 μέλη, άρα θεωρούμε ότι υπάρχει απαρτία και περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες, παρακαλώ, για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Να υπενθυμίσω στα, πολιτικά, στα μέλη ότι μια πολιτική ομάδα μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα ή τουλάχιστον τρει βουλευτέ από κοινού μπορούν να καταστάσουν μια υποψηφιότητα. Αν έχουμε λοιπόν υποψηφίου για τη θέση τη Προεδρία. Ε, να δώσω όμω πρώτα το λόγο. Α, όχι, συγγνώμη. Πριν σα δώσω το λόγο, να σα υπενθυμίσω ότι οποιοδήποτε ε, είναι υποψήφιο θα πρέπει να είναι τακτικό μέλλον, θα πρέπει να έχει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων συμπληρωμένη, να την έχει καταθέσει και τη σχετική δήλωση για την συμπεριφορά του, για την ε, δέουσα συμπεριφορά. Αν έχουμε λοιπόν υποψηφίου, για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να σα πω ότι ονομάζομαι Μπορτερ Ζόινσκα και είμαι μέλος ε, της επιτροπή Προπολογισμού. Θα ήθελα εξονόμητος του κόμματο του ECR να υποβάλλω την υποψηφιότητα του Γιώχαν Φανφέλντ για πρόεδρο της επιτροπή Προπολογισμού. Ο κύριος Φαν Όφενβελτ είναι πρώην Υπουργό Οικονομικών του Βελγίου, είναι οικονομολόγος και είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι έχει την απαραίτητη εμπειρία και τις απαραίτητες ικανότητες για να ηγηθεί της Επιτροπής. Και πραγματικά ε, θα το πράξει με άριστο τρόπο τα επόμενα χρόνια. Την υποψηφιότητα λοιπόν του κύριου Γιώχαν Φανόφερβελ θα ήθελα να καταθέσω για πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Ο κύριο Γιώχαν Φανόφερβελ κατατέθηκε ω υποψήφιο από την ομάδα του ECR των ε, συντερτικών και των Άλλοι υποψήφοι, παρακαλώ. Αν όχι, να ζητήσω από τον κύριο Φανόφερβελ κατά πόσον δέχεται την υποψηφιότητά του. Αν δέχεστε την υποψηφιότητά σας, να σας εκλέξουμε διαβοής. Γιώχαν Βαν Όφερφέλτε. Έχετε λοιπόν την Πρόεδρια τη Επιτροπή μα συγχαρητήρια και καλή τύχη σα εύχομαι. Στην εκπλήρωση των καθηκόντων σα θα σα ε, δώσω τα ίνια τη Προεδρία για να συντονίσετε την εκλογή των αντιπροέδρων. Good afternoon to you uh, all. Καλησπέρα σε όλους σας. Και καταρχάς θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ή την επανεκλογή σας. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι ιδιαίτερη η τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα σας, ε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου, τα σημαντικά καθήκοντά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ελπίζω να μπορώ να, να ελπίσω στην υποστήριξη όλων σας. Και για να είμαι απόλυτο, να σας πω πως είναι το όνομά μου είναι Γιώχαν. Γιώχαν, όχι Γιώχανα. Γιώχανα. Γιώχαν, μάλλον φαίνεται και όλο ότι είμαι Γιώχανα, αλλά εν πάση περιπτώσει το διευκρινίζω ε, και να προχωρήσουμε με τα επόμενα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Να περάσουμε με πρώτο, στην εκλογή του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου αντιπρόεδρου. Όπως επισημάνθηκε. Όσο τα πληρωματικά μέλη συμμετέχουν στην ψηφοφορία, ανακοινώθηκαν στην αρχή της συναντρίασης. Αν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή, παρακαλώ να διαβιβαστεί στη γραμματεία πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Απαρτία έχουμε. Είμαστε όσο χρειάζεται. Να υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός ε, προβλέπει να αποτυπώνεται η διαφορετικότητα του κοινοβουλίου ε, και στη σύμβαση του Προεδρείου. Άρα το Προεδρείο δεν μπορεί να παρτίζεται μόνο από γυναίκες ή άντρες. Επίσης είναι επίσης, ε, απαράδεκτο να προέρχονται όλα τα μέλη από το ίδιο κράτος μέλος. Θα θέλαμε λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου και αυτό γιατί όπως ε, σας ενημερώσαμε για τη θέση αυτή η υποψηφιότητα έχει καταθέσει μια γυναίκα. Αν συμφωνούμε λοιπόν, τουλάχιστον θα έχουμε την ε, ασφαλιστική δικλίδα ότι σεβόμαστε το κριτήριο της ισότητας των φύλων. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Υποψηφιότητε λοιπόν για την ε, τρίτη αντιπροεδρία της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Ελπίζω να συνεργαστούμε στενά για να προασπιστούμε τι θέσει του Κοινοβουλίου σε θέματα προπολογισμού εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θα ήθελα να προτείνω τη Μαργαρίτα Μάρκε για τρίτη αντιπρόεδρο. Καταρχά. να δούμε κατά πόσον είναι πλήρε μέλο, τακτικό μέλο η υποψήφια και κατά πόσον έχει ήδη ε, συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και την ε, δήλωση για την ε, δέουσα συμπεριφορά. Η κυρία Μάρκες έχει καταθέσει λοιπόν υποψηφιότητα, αν εφόσον δέχεται την υποψηφιότητά της. Φυσικά. Δέχεστε παρακαλώ την υποψηφιότητά σας, ναι βεβαίως. Τι δέχομαι. Μάλιστα διαβοής. Μιας και δεν έχουμε άλλες υποψηφιότητε. Να γίνει παρακαλώ η εκλογή. So we go from three to one. Και έτσι να περάσουμε από την τρίτη αντιπροεδρία στην πρώτη αντιπροεδρία. Okay. Sorry, just beginner's mistake. I have... Please... Τάρης είμαι, έκανα ένα λάθος. Ελάτε εδώ φυσικά στο βήμα και εσείς. Okay. So, uh, Τώρα, θέλουμε να διορίσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Κύριε Φερνάντες, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Για, τον, για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου, θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Λεβαντόφσκι. Με αυτή την ομάδα, με τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τα μέλη αυτά θα έχουμε ένα συνασπισμό υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Δέχεστε και και το, την υποψηφιότητά σας. Βεβαίω, είμαι έτοιμος για δράση. Τρεις είμαστε εδώ πέρα που είμαστε έτοιμοι για δράση, τουλάχιστον. Μπορούμε να προχωρήσουμε επίσης με την εκλογή του αντιπρόεδρου αυτού διαβοής. Κύριε Λεβαντόφσκι, ελάτε και εσείς επάνω. Και τώρα θέλω να δούμε τις υποψηφιότητες για την εκλογή του, του δεύτερου αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την ομάδα Renew Europe προτείνουμε τον κύριο Ολιβιέ Σαστέλ, που ήταν Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, και Υπουργό Προπολογισμού του Βελγίου. Κύριε Σαστέλ. Είσαστε έτοιμος να δεχτείτε την υποψηφιότητα αυτή. Πανέτοιμος. Μπορούμε να τον εκλέξουμε διαβοής. Κύριε Σαστέλ. Και τώρα θέλουμε να προχωρήσουμε στην, ε, στην υποψηφιότητα, υποψηφιότητες του τέταρτου, τέταρτου αντιπροεδρού της επιτροπη Επιτροπής. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Φερνάντες. Ο κύριος Herbst είναι η πρότασή μας. Δέχεστε την υποψηφιότητα. Μπορούμε να τον εκλέξουμε τον κύριο Herbst δια Πολύ ωραία. Θαυμάσια τα πήγαμε. Αυτό είναι ένα preview για τον τρόπο που θα εργαστεί αυτή η Επιτροπή. Από εδώ και πέρα. Τελευταία ανακοίνωση. Η ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση είναι 22 Ιουλίου, 4 ώρα το απόγευμα μέχρι 8.30 και 23 Ιουλίου, 9 το πρωί μέχρι 12.30 εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Γεια σας.